Του υποδέχθηκε η αστυνομία, του αφαιρέθηκαν τα διαβατήρια και του έστειλαν σπίτι με το πρώτο αεροπλάνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά για ευρωβουλευτές σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ακόμη περισσότερο σε μια χώρα όπως το Μαρόκο, στο οποίο, με το οποίο έχουμε φιλικές σχέσεις και με το οποίο μας συνδέουν μια σειρά έκρεμων συμβάσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω να σα ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, κατά πόσο ελήφθησαν, προβλέφθηκε κάτι για αυτό το σκοπό, να απευθυνθούμε στι Μαροκινές αρχέ για το θέμα αυτό, διότι ξέρω ότι εσεί ταξιδεύετε πολύ στον κόσμο. Πολύ συχνά έχετε έρθει και στη χώρα μου, στην Ιταλία, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση για μα. Ε, αν και εκεί ήσασταν υπό την ιδιότητά σα του αρχηγού του Σοσιαλιστικού Κόμματο αντί για πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σα ζητήσω λοιπόν να μπορέσετε να ε, παρέμβετε όσον αφορά αυτό το δυστυχέ συμβάν. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δω τι αφορούσε ακριβώς το διαδικαστικό σε σχέση με τα γεγονότα που περιγράψατε όσον αφορά την ε, αποπομπή του συναδέλφου από τις Μαροκινές Αρχές. Την προηγούμενη πέμπτη στην διάσκεψη των Προέδρων σε βάθος συζητήσαμε το θέμα η διάσκεψη των Προέδρων, τον συνάδελφο Μπρόκ υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών τον παρακάλεσε το θέμα αυτό να το εξετάσει στην Επιτροπή Εξωτερικών και να κάνει τις αναγκαίες επαφές και διαβήματα με τις μαροκινές αρχές. Και υποθέτω ότι ο κύριος Μπρόκ το έκανε ήδη. Εμένα τουλάχιστον μου είπε ότι ήδη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου ήρθε σε επαφή και συζήτησε το θέμα αυτής της περίπτωσης. Τώρα, οι αρμόδιες κυπριακές αρχές με ενημέρωσαν για τον διορισμό του συναδέφου Ιωάννη Κασουλίδη ως Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου από την 1η ε, Μαρτίου. Εξ ονόματος του Σώματος θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Κασουλίδη για τον διορισμό του ως Υπουργό Εξωτερικών της ε, Κύπρου.